Thank Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ ε, που ήρθατε και στην ε, μεικτή συνάντηση με την Επιτροπή Πολιτισμού. Ε, πια έχει γίνει παράδοση να συνεργαζόμαστε με άλλες επιτροπές, οπότε βεβαίως σε αυτές συμπεριλαμβάνουμε και την Επιτροπή Πολιτισμού. Θέλω να ξεκινήσουμε γιατί στις 12.30 ακριβώς πρέπει να σταματήσουμε τουλάχιστον τούτο το κομμάτι της ε, συνάντησης και μετά να συνεχίσουμε στις 2 η ώρα όπου θα γίνει η ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Μαριάν Τάισεν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα κάνουμε ε, μια συνεδρίαση που θα ασχοληθεί με το θέμα της απόσπασης εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και θα συζητήσουμε τις τροπολογίες Λέγοντας λοιπόν αυτό θα δώσω το λόγο στους εισηγητές και μπορείτε ε, να μοιραστείτε το χρόνο ανάμεσά σας όπως εσείς επιθυμείτε. Θα δώσουμε το λόγο λοιπόν ε, στη συνάδελφο πρώτα. Δεν ξέρω ποιος έχετε διαλέξει, ποιος θα μιλήσει πρώτος. Έχετε το λόγο, εν περιπτώσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που καταλάβατε πώς μοιραστήκαμε το φόρτο εργασίας οι Άγνες και εγώ και όπως έχουμε κάνει αρκετές φορές ήδη στο παρελθόν θα παρουσιάσουμε το σημείο αυτό για τις τροπολογίες με δύο τρόπους. Θα μοιραστούμε τα θέματα και θα σας τα παρουσιάσουμε. Και αυτό γιατί πια είμαστε πολύ συνηθισμένοι στο να συνεργαζόμαστε. Να ξεκινήσω κυρία Πρόεδρε ζητώντας συγνώμη από τους συναδέλφους, θελήσαμε να παρουσιάσουμε τις τροπολογίες τώρα, το συντομότερο δυνατόν, αλλά βέβαια δεν είναι έτοιμες ακόμα μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες. Έχουμε τα αγγλικά από τη Δευτέρα, οπότε νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα επί του οποίου μπορούμε, χρησιμοποιώντα αυτή τη μετάφραση, να εργαστούμε, σίγουρα το συντομότερο δυνατόν θα έχετε και στη γλώσσα σας το σύνολο των εγγράφων, έτσι ώστε να μπορείτε κι εσείς να δουλέψετε σε βάθος το θέμα αυτό. Ξέρουμε πως η σαφήνεια και η ακρίβεια ε, στην ορολογία εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική. Η πιο σημαντική φάση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα και τα όσα αυτή τη στιγμή μένουν να κάνουμε, ε, γιατί είμαστε απόλυτα συνδυασμένες οι Άγνες και εγώ, είναι για κάθε ομάδα, για κάθε πολιτική ομάδα, εσείς ως σκιώδης να έχετε τη δυνατότητα να παρουσιάσετε τις τροπολογίες και τις βασικούς άξονες, ε, τα όσα δηλαδή έχετε κάνει. Εμείς εδώ είμαστε οι συνεισηγήτριες και είμαστε σε φάση ακρόασης. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί σίγουρα συνεργαστήκαμε με όλους και είδαμε και τους εκπροσώπους σας, τους εθνικούς εκπροσώπους και άλλους πολλούς ακόμα. Αλλά καλό είναι ο καθένας να εκφραστεί και να πει για το σύνολο των τροπολογιών, για τους βασικούς άξονες και για τις απόψεις του, ποια είναι τα σχόλιά του. Είναι γύρω στις 500 τροπολογίες που κατατέθηκαν. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που δεν, που δεν καταθέσατε υπερβολικά πορές. Γιατί 500 ε, τροπολογίες οι οποίες για ένα κείμενο τόσο σημαντικό όπως αυτό μας λένε οι εμπειρογνώμονες πως δεν είναι και τόσες. Το καλό είναι ότι μπορούμε να τις ομαδοποιήσουμε γιατί περιστρέφονται γύρω από συγκεκριμένα θέματα. Με ανοιχτό πνεύμα λοιπόν, επειδή θέλουμε ένα πολύ ισορροπημένο κείμενο και δεν θέλουμε να υπάρχουν διαιρέσεις και θέλουμε το κείμενο αυτό να ανταποκρίνεται και στα θέματα του θεμητού ανταγωνισμού, του κοινωνικού ε, dumping, της δυναμικής που θέλουμε να δώσουμε στα θέματα απασχόλησης στην Ευρώπη. Αυτά λοιπόν, αυτές οι τροπολογίες, αυτός ο αριθμός τροπολογιών, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τις χειριστούμε ώστε να τον καλύτερα με όλες τις πολιτικές ομάδες. Και αυτές οι 500 τροπολογίες είναι μισές-μισές. Οι μισές είναι για τα εκτιμώντας και οι μισές είναι επί της ουσίας του κειμένου. Οπότε και εδώ το στοιχείο αυτό είναι πολύ σημαντικό για να το λάβουμε υπόψη μας. Ξέρετε πόσο οι ε, ουσιαστικές τροπολογίες, επί της ουσίας μάλλον, ε, είναι σημαντικές. Μπορώ να σας δώσω και τα στατιστικά αναπολιτική ομάδα, ΕΛΚ, 169, Ευχαριστώ πολύ την πολιτική μου ομάδα που έφτασε στην κορυφή του καταλόγου των όσων κατέθεσαν. Καμιά ε, εκατοντάδα οι σοσιαλιστές, Έχω τρεις πολιτικές ομάδες, ECR, Φιλελεύθερη και Γκουέ, που έχουν καταθέσει γύρω στις 50. Η Πράσινη και το EFN, ε, καμιά δεκαριά, και η DDF 7. Γι' αυτό σας τα ομαδοποίησα έτσι ώστε να ξέρετε πόσες είναι. Άγνες, θες να περάσουμε στην παρουσίαση των τροπολογιών επί της ουσίας. Εγώ μπορώ να ξεκινήσω με τη διάρκεια της απόσπασης και του εφαρμοστέου ε, δικαίου κατά τη διάρκεια αυτή. Έχουμε 110 περίπου 170 τροπολογίες νομίζω. Κάποιοι θέλουν να μην έχουμε μέγιστη διάρκεια και να παρακολουθήσουμε τα όσα έχουμε στο status quo σήμερα. Άλλοι, ε, δηλαδή τους 24 μήνες, άλλοι θέλουν 24 μήνες να αλλάξουν. Έχουμε διάφορες ε, προτάσεις, 3, 6, 12 μήνες. Κάποιοι θέλουν να υπάρχουν περίοδοι αναφοράς για τον υπολογισμό της διάρκειας και να πούμε 36 μήνες Δηλαδή εδώ έχουμε μια αύξηση και μπορούμε τη μέγιστη διάρκεια να τη συνδυάσουμε, σύμφωνα με κάποιους, με αυτό που, προ, που προτείνει το καθεστώς ε, κοινωνικής πρόνοιας μαζί με τις εξαιρέσεις που προβλέπει το κείμενο για τις ορευτικές περιόδους σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου αποσπασμένου εργαζόμενου από άλλον, πολλοί επιθυμούν να διαγραφεί η ρήτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία δεν λαμβάνει υπόψη παρά μόνο τις συμβάσεις που ξεπερνούν τους 6 μήνες. Εδώ λοιπόν μπορούμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Αυτές είναι οι βασικές γραμμές των όσων έχουν προταθεί. Γενικότερα αυτά προτείνονται για τη διάρκεια και δίνω το λόγο τώρα στην Άγνες. Ε, thank ε, ε, Σας ευχαριστώ πολύ και από τη δικιά μου πλευρά. Ευχαριστώ βέβαια και όλους τους συναδέλφους που κατέβαλαν τόσο μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να υποβάλουν τις τροπολογίες. Είμαι απολύτως πεπισμένη ότι ε, θα, ε, ότι ο καθένας μας προσπαθεί να βάλει το δικό του λιθάρι έτσι ώστε ε, πραγματικά να γίνει η καλύτερη δυνατή δουλειά. Πολλοί άνθρωποι έχουν κατεβάλει μεγάλες προσπάθειες και έχουν ασχοληθεί πολύ με το θέμα αυτό, κυρίως για τις συλλογικές συμφωνίες Για τις ε, συλλογικές ε, συμβάσεις λοιπόν όσον αφορά τους αποσπασμένους εργαζόμενους πρέπει όλοι να ε, έχουν τέτοιες συμβάσεις ανά γεωγραφική περιοχή, ανατομέα, ανα κλάδο, ανα επάγγελμα συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί από τις πιο εμβληματικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων Επίσης ε, υπάρχουν τροπολογίες ε, οι οποίες ε, προτείνουν μονάχα συμβάσεις οι οποίες να είναι καθολικές και με καθολική εφαρμογή, συλλογικές, συνολικές και με καθολική εφαρμογή λοιπόν. Για τις συλλογικές λοιπόν συμβάσεις υπάρχουν πολλές απόψεις και πολλά στοιχεία. Η αμοιβή, όσον αφορά την αμοιβή, λοιπόν, έχουμε κάποιες τροπολογίες, έχουν υποβληθεί δηλαδή κάποιες τροπολογίες, ε, οι οποίες ζητούν επιστροφή στη διατύπωση του minimum rates of pay και όχι ε, αμοιβή, να μην γίνεται πλέον λόγος για αμοιβή, αλλά για ελάχιστο ε, μισθό. Πρέπει να σας πω ότι η αμοιβή είναι ο ελάχιστος μισθός και τα επιδόματα τα οποία ε, μπορούν να υπάρξουν. Είτε είναι επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών, είτε οποιοδήποτε άλλο επίδομα. και ορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε οι εθνικοί εργαζόμενοι και οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι της χώρας υποδοχής ε, να ε, μην έχουν διαφορετική αντιμετώπιση έτσι ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε ε, αθέμητος ανταγωνισμός είτε οποιαδήποτε πρόβλημα ας πούμε αθέμητων κοινωνικών σχέσεων. Αυτό όσον αφορά το θέμα της αμοιβή. Επίσης, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες, 23 αν δεν κάνω λάθος, οι οποίες θέλουν να καθορίσουν ποιο είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό τη αμοιβή. Σας μιλώ ειλικρινά και πρέπει να σας πω ότι η σκέψη των δύο συνεισηγητριών και το μέλημά τους είναι να ενεργήσουν έτσι ώστε να γίνει σεβαστή η έννοια της αμοιβή που θα καθορίζεται από το κράτος μέλος. Δεν πρέπει η Ευρώπη να, παρεμβαίνει, να συγγνώμη, στον καθορισμό αυτής της αμοιβή. Υπάρχουν δύο τροπολογίες, δύο τροπολογίες, αναφέρουν μια ιδέα που είχε αναφερθεί από την ε, Σλοβακική Προεδρία στο Συμβούλιο με ναι, τον ορισμό ενός συστήματος περίπλοκου που ε, ε, αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρξει μία πρώτη περίοδος 6 μηνών και μετά 26, ε, 24 μηνών, δηλαδή από 6 μέχρι 24 μήνες και μετά από τους 24 μήνες και εφεξής ένα άλλο καθεστώς. Τρία καθεστώτα δηλαδή, μέχρι 6 μήνες, από 6 μέχρι 24 και πέραν των 24. Πρέπει να σας πω ότι εγκατελείφθη στο Συμβούλιο η άποψη αυτή και δεν συζητιέται καν πλέον και επομένως ίσως καλό θα ήταν οι συγγραφή ε, αυτών των ε, τροπολογιών να μας εξηγήσουν ακριβώς ε, τι εννοούν και τι θα ήθελαν. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά και οι Αγνές και εγώ η ίδια πιστεύουμε ότι καλό θα ήταν να έχουμε συστήματα απλά όσον αφορά τη διοίκηση και σαφή όσον αφορά τον έλεγχο. Στρέφουμε προς την Τζανούτα η οποία ασχολήθηκε με τον κανονισμό ελέγχου των αποσπασμένων εργαζόμενων και επαναλαμβάνω ότι το κείμενό μας θα πρέπει να είναι σωστό και θα πρέπει να είναι συνεκτικό και συντονισμένο με το κείμενο για τους ελέγχους. Όσο πιο περίπλοκα κάνουμε τα πράγματα, τόσο λιγότερο θα πετύχουμε μια καλή εφαρμογή. Υπάρχουν επίσης κάποιες τροπολογίες για, το, για την ιστοσελίδα στην οποία θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αναφέρουν όλες τις ε, πληροφορίες σχετικά με τις ε, συμβάσεις κτλ. Ε, με τον τρόπο αυτό ε, μπορεί να προσθεθεί ο έλεγχος ή τα στοιχεία των αποσπασμένων εργαζομένων και θα διευκολύνει επίσης και την εργασία, το, το έργο μάλλον των επιχειρήσεων που θα ξέρουν πλέον και των εταιριών που θα ξέρουν πλέον τι πρέπει να σεβαστούν. Ναι, ίσως όμως πρώτα να μιλήσουμε για, τα, για τις δαπάνες και τις απαλλαγές ορισμένων ή τις κάποιες μειώσεις από τους μισθούς. Αυτό είναι το ένα. Μετά πρέπει να μιλήσουμε βέβαια και για τις υπεργολαβίες. Καταρχάς δαπάνες. Και υπολογισμός κάποιων δαπανών ως μείωση των μισθών γιατί κάποιοι λένε ότι θέλουν να βάλουν εθνικούς κανόνες ως προς την καταβολή δαπανών για, το, για ταξίδια, για στέγη, διαμονή καλύτερα, ως επιπλέον επιβάρυνση για τον αποσπασμένο, στον ορισμό δηλαδή της αμοιβή. Αυτή την προσθήκη λοιπόν τη συνοδεύουν οι συνάδελφοι με το σχόλιο ότι αυτές οι δαπάνες δεν μπορούν να αφαιρεθούν από το μισθό ή ότι δεν μπορεί να υπάρξουν άλλες ε, μειώσεις στον υπολογισμό, άλλες εκπτώσεις θα λέγαμε, ε, από ε, κατάρτιση και άλλα μαθήματα. Δηλαδή πρέπει να είναι ευρύτερη η έννοια της αμοιβή. Θα υπολογίζονται και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής αλλά και εξοπλισμού, κατάρτισης κτλ. Ταυτόχρονα ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν υποστηρίζουν την πρόταση αυτή. Πρέπει να διατυπώσουμε όμως το τελικό κείμενο της πρότασής μας και ως εκ τούτου επανέρχομαι στην ε, σχετική και με τις συλλογικέ συμβάσεις ε, πρόταση, με την επιλογή της λύσης για τις συλλογικέ συμβάσεις, πρόταση των, ε, για την απόσπαση. Εδώ υπάρχουν πολλές τροπολογίες που στοχεύουν στον τροποποίηση ή και κατάργηση της πρότασης Επιτροπής. Θα θυμάστε ότι η Επιτροπή είχε υπενθυμίσει ότι αν υπάρχει εθνική υποχρέωση για τους υπεργολάβους, αυτή η δέσμευση θα πρέπει να ισχύει και για τον αποσπασμένο εργαζόμενο. Και άρα θα έπρεπε αυτές οι δεσμεύσεις να ενσωματώνονται και να εγγράφονται σε μία συλλογική σύμβαση επίπεδου επιχειρήσεως που θα ισχύει και για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Επομένως, εκεί λύνεται το ζήτημα της απόσπασης και της υπεργολαβίας. Κάποιοι συνάλφοι υποστηρίζουν με τις τροπολογίες τους την ιδέα αυτή. Κάποιες άλλες τροπολογίες όμως την απορρίπτουν και λένε ότι δεν πρέπει ποτέ σε επίπεδο επιχειρήσεως μια συλλογική σύμβαση ε, επιχειρησιακή να, ε, να ισχύει και για τους αποσπασμένους. Η Ελίζαμπετ τώρα για την ε, κάλυψη της διαμονής. Θα είμαι απόλυτα σαφής. Υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες που προτείνουν να υποστηρίξουν αυτό που είχαμε εμείς ε, προτείνει με την έκθεσή μας, το σεβασμό δηλαδή των καλών συνθήκων διαμονής, κάτι το οποίο μας βοηθάει και για τη συνέχεια. Ούτε βέβαια μας ξαφνιάζει το ότι υπάρχει αυτή η υποστήριξη, γιατί ξέρουμε ότι όλε οι πολιτικέ ομάδε που συμμετέχουν στην Επιτροπή μα υποστήριζουν τι ιδέε αυτέ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ τώρα περνώ στο τελευταίο διπλή απόσπαση και ε, εταιρείε γραμματοθυρίδες. Υπάρχουν κάποιες ε, τροπολογίες αρκετές οι οποίες έχουν ε, να κάνουν με το λεγόμενο generic posting και την αντιμετώπιση του, ε, με το genuine posting, συγγνώμη, ε, γνήσια απόσπαση, ότι δηλαδή εάν δεν είναι γνήσια η απόσταση, απόσπαση, λένε κάποιες τροπολογίες, από την πρώτη μέρα πρέπει να ισχύει η νομοθεσία της χώρας υποδοχής, εκτός και αν ευνοϊκότεροι η όρη στη χώρα ε, προέλευσης, ενώ κάποιες άλλες τροπολογίες είναι κάπου, είναι λιγότερο αυστηρές, μιλούν για υπολογισμό του κύκλου εργασιών, του υπεργολάβου που αποσπά σε άλλη χώρα, στη χώρα εγκατάσταση, στη χώρα έδρας, ή περιορισμό στο ποιου εργαζόμενου, πόσου εργαζόμενου μπορεί να αποσπά ή ποια μπορεί να θεωρήσει την έδρα ή την, ε, τον τόπο μόνιμη κατοικία των εργαζομένων αυτών. Ορίζεται πάντως μια ελάχιστη περίοδος για την οποία ο αποσπασμένος εργαζόμενος πρέπει να έχει ε, εργαστεί πριν να ε, αποσπαστεί και να υπαχθεί στην λύση αυτή. Άλλες τροπολογίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις καταχρήσεις, τις καταστρατηγήσεις. Λένε ότι δεν μπορεί η απόσπαση να αφορά δύο διαφορετικές δικαιοδοσίες ή εάν αφορά πάνω από δύο δικαιοδοσίες, τότε αυτομάτως ισχύει τον δίκαιο της χώρας υποδοχής, εκτός και αν η χώρα προελεύσεω έχει ευνοϊκότερε ε, διατάξεις. Επίσης κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζονται νέοι κανόνες, αλλά ότι η λύση θα δοθεί μέσω της καλύτερης εφαρμογής και επιβολής της ισχύουσας νομοθεσίας από τις εθνικές αρχές και δει άρθρα 3 και 4 της οδηγίας περί ε, εφαρμογή στις οδηγίες αυτής που έχει τεθεί εντωμεταξύ ενισχύ Η άποψή μου, αλλά και της Ελίσσαπετ, είναι ότι και η καλύτερη εφαρμογή και οι καλύτεροι κανόνες μπορούν να προχωρήσουν και πρέπει να προχωρήσουν χέρι-χέρι. Και αυτή είναι η θέση στην οποία, την οποία χρησιμοποιούμε ως βάση εργασίας. Αυτά από μένα προς το παρόν. Περιμένουμε να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Ευχαριστώ και δύο λόγια ακόμα για την απόσπαση από εταιρείε προσωρινής απασχόλησης, interim. Μια πρόταση υπάρχει σχετική με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής με αυτές τις ε, ε, υπηρεσίες, τις εταιρείε. Άλλες τροπολογίες δεν φτάνουν μέχρι εκεί, αλλά λένε ότι θα πρέπει κάποιες ε, συγκεκριμένες περιστάσεις να περιγραφούν με στην νομοθεσία, ενώ κάποιοι βουλευτές έχουν καταθέσει τροπολογίες σχετικές με την εισαγωγή της 3, του άρθρου 3 παράγραφος 9 που προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσει και που είναι πιο αυστηρό από αυτό της Επιτροπής ε, γιατί βλέπουμε ότι αυτό ακολουθεί και το πνεύμα των προτάσεών μας. Επομένως μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, να ακούσουμε τα δικά σας επιχειρήματα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μάκιντάιερ, ECR, Σιώδης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες για τα όσα έχουν κάνει μέχρι τώρα. Γνωρίζω πως σε προηγούμενες ανταλλαγές απόψεων έχω ήδη συζητήσει για μια σειρά από και πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να μην φέρουμε τη διαίρεση στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι κάποιες από τις τροπολογίες οι οποίες έχουν υποβληθεί δείχνουν ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση στις απόψεις μας και νομίζω ότι καλό θα ήταν ε, να μην διαιρούμε την Ευρώπη ε, σε ανατολική και δυτική. Νομίζω πως για να βρεθεί μια συνενετική λύση θα πρέπει να κάνουμε πολύ δρόμο και να βρούμε κάποιες λύσεις που στην πράξη θα λειτουργήσουν και για όλα τα κράτη-μέλη και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους. Οπότε δεν είναι που εκτιμώ ε, το σύνολο της εργασίας που ακόμα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει καταρχήν να κλείσουμε τα παραθυράκια που ε, επιτρέπουν τις ψευδοαποσπάσεις και να δούμε και τη διάσταση προστασίας των εργαζομένων. Αλλά δεν θέλω καθόλου μέτρα που είναι προστατευτικά. Και νομίζω ότι κάποιες χώρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ενδεχομένως κάποιους από αυτούς τους κανόνες ως ε, προστατευτικό μέτρο, κάτι το οποίο θα έβρισκα ιδιαίτερα λυπηρό. Φοβάμαι πως αντίθετα με τα όσα είπε μόλις οι Άγνες, πιστεύω πως θα πρέπει όντως να εστιάσουμε στην εφαρμογή των ε, τριχών των κανόνων πριν κάνουμε ριζικές αλλαγές σε κάτι το οποίο είναι ένα τοπίο ε, νομοθετικά μιλώντας, εξαιρετικά σύνθετο. Έχω και δύο πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Δηλαδή, μακροπρόθεσμες αποσπάσεις που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις όταν στέλνουν εργαζομένους σε κάποια, κάποιο παράρτημά τους ε, σε άλλη χώρα, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να μείνουν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις αυτές να έχουν τη δυνατότητα της ευελιξίας που να τους επιτρέπει αυτή η δουλειά να γίνεται εύκολα και ελπίζω οι εισηγήτριες να αντιμετωπίσουν με θετικό πνεύμα τις τροπολογίες μας ε, σχετικά. Το άλλο που ήθελα να συζητήσω είναι πώς θα καταλάβουμε και πώς θα κατανοήσουμε ε, πώς εργάζεται ο κόσμος πια σήμερα. Δηλαδή, οι βιομηχανίες δεν πολλούν απλώς προϊόντα. Όχι. Ένα ολόκληρο πακέτο υπηρεσιών που πλησιώνει τα προϊόντα αυτά πολλούν. Και θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τη Μαρτίνα, γιατί σήμερα το πρωί ε, στο πρωινό γεύμα ε, κάνουμε μια συνάντηση με τις επιχειρήσεις, οι οποίες μας είπαν πόσο δύσκολο είναι όταν προσπαθούν να φτιάξουν ένα μηχάνημα. Δηλαδή, ε, στη σύμβαση λέει ότι εκτός από το μηχάνημα πρέπει να αναλάβουν και τις συντήρηση του μηχανήματος και αυτό πρέπει να γίνει σε χρόνο ρεκόρ. Δεν έχουν το χρόνο να ζητήσουν, να αιτηθούν, να καταχωρηθούν, να συμπληρώσουν αιτήσει και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως υπάρχει αυτός ο νέος τρόπος εργασίας. Thank you. Uh, I'll give the floor to... Η κυρία Γκλαβαγιώβα είναι η επόμενη ομιλήτρια και σας ζητώ να είμαστε όλοι σύντομοι γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Είναι δύσκολο να είναι κανείς σύντομος εάν θέλει κανείς να ε, λάβει υπόψη όλα τα θέματα. Νομίζω πως ο δρόμος μπροστά μας θα είναι μακρύς, είναι 500 ε, τροπολογίες που δείχνει πως είναι και σημαντικό το θέμα αλλά είναι και ε, όπως είπατε και εσείς, πηγή διαιρέσεων. Δεν θα μιλούσα τόσο πολύ για την ποσότητα, αλλά για την ποιότητα των τροπολογιών, γιατί νομίζω ότι εδώ αντιμετωπίζουμε τις βασικές, τα βασικά ζητήματα που έχουμε ακούσει και στο παρελθόν κατά την ανταλλαγή απόψεων. Επειδή δεν έχουν συναντηθεί οι σκιώδες καθόλου, σας ζητώ δημόσια εσείς τις να λάβετε υπόψη όλε τι φωνές που ακούστηκαν, να τι αξιολογήσετε σε βάθος και να προτείνετε συμβιβαστικές λύσεις οι οποίες θα ξεπερνούν την, ε, το εθνικό πολιτικό τοπίο, γιατί νομίζω πως αυτή τη στιγμή χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Ελπίζω πως πολλές αντιστροπολογίες θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο ε, συμβιβασμού και θα ήθελα να βασιστούν οι δικές μας τροπολογίες στα στοιχεία, στα δεδομένα, στην υπάρχουσα νομολογία και να είμαστε σίγουροι πως αυτό που κάνουμε είναι ρεαλιστικό για όσους προχωρούν σε απόσπαση εργαζομένων. Και γι' αυτό ε, οργάνωσα αυτό το πρωινό σήμερα. Ήθελα να μας πούνε οι επιχειρήσεις την πραγματικότητα τι γίνεται, ποιες είναι οι πραγματικές προκλήσεις και τα προβλήματα. Και στα σύντομα θα αναφερθώ σε τέσσερα σημεία γιατί ξέρετε τι είναι αυτό που με ανησυχεί. Πρώτον, η διάρκεια. Ακόμα αμφιβάλλω για το ότι πρέπει να θέσουμε οποιονδήποτε περιορισμό, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι σημαίνει η, απόσπαση, αν είναι πραγματική ή όχι. Ε, γιατί εκεί βρίσκεται το όλο θέμα. Όχι ο περιορισμό σε διάρκεια, αλλά η αυθεντικότητα της απόσπασης. Επίσης, οι αμοιβέ είναι προφανές πως κάποιοι ευρωβουλευτές οι οποίοι είναι από χώρε που υπάρχει ελάχιστο, ε, ελάχιστος μισθός θέλουν να ακολουθήσουμε τη διατύπωση που λέει minimum rates of pay. Εντάξει, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό. Μετά, α, υποεργολαβίες. Ζήτησα να διαγραφεί αυτή η υποχρέωση, γιατί αν γίνεται υπεργολαβία είναι ασαφές α, πώς και τι. Άρα λοιπόν καλό είναι, υπάρχει κοινή πρόθεση αυτό το κομμάτι να διαγραφεί. Επίσης, μεταφορές. Δεν μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί το θέμα εδώ με αυτή την νομοθεσία. Περιμένουμε τώρα την πρόταση ε, από την Επίτροπο Μπούλτς, η οποία μας είπε πως θα έχουμε ε, συγκεκριμένη νομοθεσία για τον κλάδο των μεταφορών, οπότε θα πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη. Διαφορετικά δεν ξέρω τι θα κάνουμε, είναι πολύ ευαίσθητο. Τέλος να σας πω πως επιμένω, επιμένω στο να είναι σαφείς οι κανόνες, ε, απλοί για τις επιχειρήσεις, και να μην επιβάλλουμε υπερβολική γραφειοκρατία σε επιχειρήσεις. Όλοι θα ευνοηθούμε από την απόσπαση των εργαζομένων. Και νομίζω ότι οι οικονομίες όλων μας θα αναπτυχθούν ε, λόγω ακριβώς αυτής της απόσπασης που έχει λάβει η χώρα σε προηγούμενα χρόνια. Θέλουμε κινητικότητα λοιπόν που να την εξασφαλίσουμε και για τις επόμενες γενιές και να σας πω πως αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Οπότε ε, με χαρά θα συνεργαστώ μαζί σας και νομίζω σε πολύ ε, εντατικές ε, συναντήσεις των σκιωδών. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Κύριε Κάρη, πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς και πάλι τις εισηγήτριες. Πολύ καλή η συνεργασία. Ανοιχτό πνεύμα συνεργασίας, είχαμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε τις τροπολογίες. Είχαμε πολλές τροπολογίες λοιπόν και ε, προσπαθούμε να τις αξιολογήσουμε με βάση ένα σημείο κίνησης που είναι και το θεμελιωδέστερο, να εξασφαλίσουμε ισότιμο επίπεδο αμοιβή για την ίδια δουλειά στην ίδια θέση. Αυτή είναι η βάση της ε, θεώρησής μας, όπως είχε πει και ο κύριος Γιούνκερ. Αυτό λοιπόν είναι η βάση, είναι άλλωστε ανεγνωρισμένο και παραδεδεγμένο. Ταυτόχρονα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και μεγάλες διαφορές μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών σε σχέση με την νομοθεσία που αφορά εθνικές συμβάσεις, τοπικού χαρακτήρα, διαφορές που υπάρχουν σε διάφορα επίπεδα, γεωγραφικά και τομεακά και πρέπει να τις λάβουμε υπόψη. Τώρα εμείς εξετάζουμε αυτήν την δυνατότητα, αυτή τη διαφορά, έτσι ώστε να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο κάποιες επιχειρήσεις να ποντάρουν και να αντλήσουν όφελος αξιοποιώντας εκείνους που βρίσκονται στις δυσμενέστερες συνθήκες. Και έτσι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν η δυνατότητα για τοπικού, τοπικής εμβέλειας συμβάσεις ή τομεακής ή κλαδικής. Ε, επίσης, Πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα της αμοιβή. Πρέπει να έχουν το δικαίωμα ή ε, κοινωνικοί εταίροι, εάν θεωρούν σκόπιμο, να ορίσουν μόνοι τους τις αμοιβέ σε ψηλότερο επίπεδο. Επίσης, θα πρέπει η απόσπαση να έχει χαρακτήρα προσωρινό, περιορισμένο χρονικά. Δεν αποκλείεται κάποιο να θέλει να πιάσει σε μια άλλη χώρα για να εργαστεί. Αλλά αν πρόκειται για απόσπαση πρέπει να είναι γνήσια απόσπαση με τα χαρακτηριστικά και του περιορισμού του χρονικού. Και αυτό για να ικανοποιούνται και οι όροι της προστασίας των δικαιωμάτων. Θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι ώστε να ε, αποτρέπεται η δραστηριοποίηση εικονικών ε, εταιριών, επιχειρήσεων και αυτές ήταν είναι οι δικές μας θέσεις. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και του εισηγήτρες και του συνεισηγητές που έχουν καταθέσει τις τροπολογίες τους. Βλέπω βεβαίως ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των θέσεών μας όλων, ότι έχουμε τις αποκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα από τις τροπολογίες αυτές εγώ διαβάζω ότι θέλουμε όλοι να εργαστούμε και να συνεργαστούμε για να βρούμε μια καλή λύση που και θα διευκολύνει την απόσπαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και θα εξασφαλίσει προστασία των δικαιωμάτων. Μια καλή κοινή θέση, μια ισχυρή κοινή θέση πάνω που όλα πρέπει να επιδιώξουμε όλοι. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι οι τροπολογίες έχουν συνταχθεί σε πνεύμα ε, που γνώμονά του έχει το όφελος όλων των Ευρωπαίων, όλων των Ευρωπαίων και εκείνων που θα πάνε να εργαστούν σε ένα άλλο κράτος μέλος, αλλά και εκείνων που μένουν στη χώρα τους και εργάζονται σε αυτή, ώστε να μην φέρουμε τους μεν αντιμέτωπους με τους δε, αλλά να εξασφαλίσουμε μια ε, κατάσταση που θα είναι υποφελής για όλους τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα επιμείνω σε κάποια σημεία που τόνισαν ήδη οι συνάδελφοι νωρίτερα. Καταρχάς για μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει νομική βάση και να μην ε, περιοριστούμε σε μια νομική βάση που αφορά μόνο την ελευθερία ε, παροχής υπηρεσιών αλλά και, τα, και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά και την ελευθερία της διακίνησης των εργαζομένων γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να αντανακλάται στη νομική βάση της ε, πρότασης. Στις αμοιβέ θα πρέπει να υπάρξει επέκταση και αυτό όμως το καταγράφεται στις τροπολογίες μας η έκπτωση από τον υπολογισμό των εξόδων κατοικίας και ε, διαμονής και ταξιδίου ε, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει διτά να αναφέρεται στην οδηγία ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να αφαιρεθούν από τον υπολογισμό αυτά. Επίσης, προσωρινή πρέπει να είναι πάντοτε η απόσπαση, το λέμε αυτό υπάρχει στο τωρινό κείμενο και πρέπει να παραμείνει η αναφορά και να είναι σαφής ο ορισμός του τι σημαίνει προσωρινή, προσωρινός ε, χρόνος για την απόσπαση. Θα το συζητήσουμε και στους συντονιστές. Επίσης, οι συλλογικέ συμβάσεις. Είναι πάρα πολύ περιορισμένος ο αριθμός των συλλογικών συμβάσεων που καλύπτουν τους ε, αποσπασμένους εργαζομένους. Στη Γερμανία, επί παραδείγματι, 17.000 συλλογικέ συμβάσεις έχουμε, εκ των οποίων μόνο 20 ισχύουν για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Γι' αυτό, λοιπόν, θα συμφωνήσετε, πιστεύω ότι πρέπει να επεκταθεί το πεδίο ε, κάλυψης και των συλλογικών συμβάσεων. Βεβαίως είναι διαφορετικά, διαφορετικές νομικές παραδόσεις και πρακτικές ε, στα κράτη-μέλη και πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία θα καλύπτει όλες τις χώρες, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ταυτόχρονα μια, μια τόσο μεγάλη απόκληση ως προς την εφαρμογή των συλλογικών ε, συμβάσεων και στους πεσπασμένους εργαζομένους από κράτος σε κράτος. Ναι, Πρόεδρε, τελειώνω. Θα πρέπει να παρεμποδίσουμε βέβαια την καταστρατήγηση ε, μέσω μη γνήσιας απόσπασης των διατάξεων. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ αυστηροί προς τη γνησιότητα της απόσπασης. Ο χώρος των μεταφορών είναι αυτός ο οποίος έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα και οπωσδήποτε πρέπει να συμπεριληφθεί ώστε να ισχύσει η οδηγία και στις μεταφορές. 30 μόνο τροπολογίες έχουμε καταθέσει, το ανέφερε και η Ελιζαμπέτ. Και αυτό γίνεται γιατί θέλουμε να αποδείξουμε ότι ως πράσινοι και έχουμε συνε... συνεπεί, συνεπείς θέσεις στην υπόθεση αυτή, αλλά και θέλουμε να συνεργαστούμε με τις άλλες πολιτικές ομάδες για να βρούμε λύσεις. Στη συνεδρία των σκιο... Η συνεδρία των Σκιωδών ήταν μια πρώτη, ένα πρώτο στάδιο μόνο. Ε, μετά από αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ακολουθούν τα στάδια της επικοινωνίας και της διαπραγμάτευσης με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε στο δυνατόν πιο γερή θέση εκ μέρους του Κοινοβουλίου για την περαιτέρω διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ. Η Λάουρα δεν είναι εδώ. Ο κύριος Μαρτάν, επομένως, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δεν θα εκπλαγείτε αν σας πω ότι προβληματιζόμαστε ενοχλούμαστε από αυτήν την εργασία στο και αν πρέπει να λάβει χώρα, διότι εμείς θέλουμε να καταρθεί με μία κοντιλιά αυτό το θέμα των αποσπασμένων εργαζομένων. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι θεωρούμε ότι ε, το κοινωνικό dumping που βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, προέρχεται ε, ε εν πολλής από, από αυτή την δυνατότητα και δεύτερον ότι αυτά που γίνονται είναι ψηλομασκαρέματα, δεν πρόκειται να τροποποιήσουν σημαντικά το θέμα. Ε, μάλιστα η κυρία Τακνού πολύ καλά το ε, ανέφερε. Είπε ότι το θέμα είπε ότι είναι στην ουσία ανταγωνισμό ανάμεσα στι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη και στι χώρε τη Δυτική. Και βεβαίω οι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη τα πάντα μπορούν να κερδίσουν και γι' αυτό επιμένουν να ε, εξακολουθήσει να ισχύει αυτή η οδηγία. Οι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη επίση ε, βεβαίω ενδιαφέρονται να συνεχίσει η ισχύ της οδηγίας αυτής γιατί έτσι κερδίζουν χρήμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν με υπεργολαβία βεβαίως θέλουν γιατί μπορούν είτε να χρησιμοποιήσουν αυτά, τις δυνατότητες που τους δίνει η οδηγία αυτή είτε να κηρύξουν πρόκειται και να κλείσουν το μαγαζί ε, και ε, Επίσης, ε, γενικότερα επιχειρήσεις, το μόνο που τους ενδιαφέρει ε, είναι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις ε, ενδιαφέρονται γιατί με τον τρόπο αυτό μειώνουν τον όγκο τον μισθολογικό και επομένως δίνουν χαμόγελα περισσότερα στους αμετόχους Οι δύο εισηγήτριες λοιπόν, μία εκ των οποίων έχει δύσκολο όνομα, αναφέρθηκαν ε, στα θέματα, μας είπαν ε, τις τροπολογίες ε, οι οποίες υπάρχουν. Το ζήτημα είναι, λένε, ότι θα πρέπει να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο το κοινωνικό dumping και να προστατέψουμε λοιπόν τους ε, δικούς μας εργαζόμενους, εθνικούς εργαζόμενους. Αυτές, αυτοί είναι δύο μεγάλοι στόχοι για μας. Εμείς λέμε ότι διατηρώντας την ε, οδηγία, ε, αφού πρέπει, θα πρέπει να υπάρξει ενορμάνωση, εναρμόνιση συγγνώμη, των ε, ε, νόμων που ισχύουν ε, στην χώρα από την οποία προέρχεται ο εργαζόμενος και στην χώρα υποδοχής και με τον τρόπο αυτό θα βρεθεί κάποια ισορροπία ανάμεσα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ε, ε, δεν έχουμε. Μία ώριτσα έχουμε ακόμα. Επομένω πρέπει να κλείσει ο κατάλογο και επομένω θα πρέπει και οι δύο εισηγήτριε, η κυρία Μωρέν Σαρτιέ και η κυρία Σάλτερ Μόζε, ε, να ε, μπορέσουν να πάρουν το λόγο. Mr. Lenners, it's Mr. Kukan, it's Thomas Mann, it's Danuta Jasloweka, it's eh, Renate Weber, uh, eh, Madam Schroederova, Helga Stevens, and then uh, hopefully Ole Christiansen, uh, and then Uh, the rapporteurs, and then we close the list. That means that you will not be able to speak three minutes as has been allowed. Λοιπόν, ε, ε, να προσέχετε να μην ξεπεράσετε τον χρόνο σας και η Χέλγκα Στίγεβενς είναι. Ναι, κοιτάξτε, εγώ είμαι, εγώ είμαι σκιώδης και Α, εγώ είμαι σκιώδης και επομένω, γιατί με βάλατε στους τελευταίους ομιλητές. Πρέπει να έχω τον κανονικό μου χρόνο ομιλίας. Ναι, αλλά η κυρία Μακεντάιερ μίλησε εξ ονόματο της ομάδας σα ε, και εξ ονόματο των σκιωδών. Θα πω κι εγώ δύο λόγια. Για μία ακόμα φορά Για μία ακόμα φορά θα ήθελα ε, να ε, πω ότι βεβαίως ε, είναι ενδιαφέρουσα αυτή η δυνατότητα για τους εργαζόμενους, για το συνάλλαγμα κτλ. Αλλά θα πρέπει η νομική βάση να σχετίζεται και με την ενιαία αγορά. Αυτό είναι προφανές. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη διάφορες αποφάσεις δικαστηρίου, ιδιαίτερος δε ε, η απόφαση για την ε, υπόθεση Λαβάλ και κυρίως θα πρέπει να λυθεί το θέμα των μεταφορών, στον τομέα των μεταφορών που έχουμε τα περισσότερα προβλήματα. Επίσης, ε, αρμοδιότητα για, την, για την, το μισθό, για την αμοιβή έχουν μόνο τα κράτη-μέλη και έτσι θα πρέπει να μείνει και η Ευρώπη δεν είναι δυνατόν όμως να δεχτεί αυτό ε, το dumping των μισθών και την διαρκή ε, ε, χειροτέρευση των συνθήκων επιτόπου. Εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να οριστούν συγκεκριμένα χρονικά όρια γιατί έτσι θα μπερδευτούν ακόμα περισσότερο και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. και εν πάση περιπτώσει όμως θα πρέπει να δούμε γιατί μετά από 24 μήνες θεωρούνται ακόμα ε, οι εργαζόμενοι αποσπασμένοι. Ε, αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τη δυνατότητα να αναλυφθεί δράση άμεσα. Ε, αυτά ήθελα να πω και κατά αυτή την έννοια υπέβαλα τροπολογίες και θα δώσω τον λόγο τώρα στον κύριο Πάβελα. Και να μην κολλησιεργούμε, έχουμε λίγο χρόνο. Θα μιλήσω γερμανικά. Βεβαίως, τα νέα κράτη-μέλη έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την οδηγία αυτή. Ξεκινώ με ερωτήματα καταρχάς. Που μερικές φορές με κρατάνε άγρυπνο. Πώς θα κάνουμε στην πράξη τη διατύπωση των τροπολογιών μας και πώς θα ε, διαμορφωθούν οι συνέπειες από τις τροπολογίες αυτές για εκείνους που ήδη εργάζονται αποσπασμένοι με βάση το παλαιό καθεστώς. Αυτό είναι το κριτήριο και ο γνώμονας για μένα. Και θα ήθελα να μου δώσουν εξηγήσει οι, οι συγγήτριες. Αν κάποιος δεν σέβεται όμως τους κανόνες που ισχύουν, δεν τους στηρεί. Με αυτούς τους νέους κανόνες θα ενθαρρυνθεί να σέβεται την νομοθεσία. Η δική μου απάντηση είναι όχι, γιατί δεν του ενδιαφέρει τι αποφασίζουμε εδώ. Οι εταιρείε ταχυδρομικές θηρίδες. Εδώ ε, συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να τις πατάξουμε πάρα πολύ αυστηρά. Μια άλλη, ωστόσο, πτυχή είναι ότι μπορεί μια οδηγία να έχει διατάξει τόσο αυστηρέ μέσα που να οδηγήσει σε μόνιμη αποδημία εργατικού δυναμικού. Τι θα γίνει για τις χώρες οι οποίες θα μένουν χωρίς εργατικό δυναμικό. Ή η διάταξη περί απόσπασης εργαζομένου που έχει ήδη ένα παρελθόν στην επιχείρηση. Ε, πώς θα προσλάβει νέο προσωπικό τότε ή τι θα κάνει με το νέο προσωπικό η εταιρεία ο υπολογισμός στο μισθό των δαπανών, ε, του επιδόματος ε, Χριστουγέννων κτλ. Αυτά πώς θα υπολογιστούν αν κάποιος δουλεύει μόνο για έξι μήνες. Θα παίρνει το ένα δεύτερο ε, ή έξι δωδέκατα του επιδόματος. Θα υπάρχει κάποιος τρόπος υπολογισμού, θα το παίρνει ολόκληρο. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω ότι εδώ πέρα ό,τι και να κάνουμε θα ισχύσει μόνο ή θα αφορά μόνο αυτούς οι οποίοι τηρούν την νομοθεσία. Από αυτά που ακούσαμε λοιπόν, ε, μπορώ να συμφωνήσω με πολλά από αυτά που είπε η θα αφορα μονο αυτού αλλά δεν μπορώ να δεχθώ αλλα δεν μπορω να δεχθω ενα τον περιορισμό στο εξάμεινο της διάρκειας. Ευχαριστώ, κύριο Κώστα έχει το λόγο. Σας παρακαλώ Πρέπει να είστε πολύ σύντομο. Η κυρία, ε, ο κύριο Κώσσα. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, με όλο το σεβασμό που έχω για σας, ε, για σας αγαπητές ε, συνείγοι συγγήτριες, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά έχετε κάνει καταπληκτική δουλειά. Δεν έχω πιστεί ακόμα πως η όλη διαδικασία είναι απαραίτητη. Εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε με αυτά που έχουμε μπροστά μα να καταφέρουμε το καλύτερο. Είναι ένα θέμα το οποίο έχω θέσει ε, πάρα πολλέ φορές, γιατί δεν νομίζω ότι ε, εδώ μιλάμε για οποιαδήποτε αντιπαράθεση μεταξύ Ανατολική και Δυτική Ευρώπη. Πρέπει να σα πω πω. Ε, ε, πως ε, η αρχή της ε, ίσης αμοιβή και ίσης εργασίας θα πρέπει θα πρέπει και σε τοπικό επίπεδο να εφαρμοστεί και όχι μόνο όταν μιλάμε για απόσπαση εργαζομένων. Και μόνο τότε θα έχουμε την αξιοπιστία να μπορούμε αυτό να το, να το μεταφέρουμε και σε άλλα κράτη-μέλη. Και αναφέρουμε στη Γερμανία, η οποία θα πρέπει πρώτη να κάνει αυτή την προσπάθεια. Να σας πω πως οι συμβασιούχοι αυτή τη στιγμή αμείβονται με χαμηλότερες αμοιβέ από τους μονίμους υπαλλήλους κάποιων εταιριών. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει και στην περίπτωση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου οι contract agents αμείβονται χαμηλότερα από τους υπαλλήλους και όταν έγραψα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μου απάντησαν ότι ξέρετε είναι διαφορετική όρη κτλ. Άρα λοιπόν για την νομική βάση ε, να σας πω ότι υπάρχει αυτό το θέμα και επίσης είμαι πεπισμένος πως εδώ αυτά τα προσπαθούμε να κάνουμε είναι η λάθος ε, προσέγγιση ε, και θα πρέπει να, κάνουμε, να, να ακολουθήσουμε διαφορετικό σκεπτικό. Θα πρέπει τους εργαζομένους να τους ε, προστατεύουμε, γιατί βέβαια διακυβεύεται εδώ και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Λοιπόν, μην ξεχνάμε πως έχουμε τον κανονισμό Ρώμη 1, και αυτός ο κανονισμός θα πρέπει να αναθεωρηθεί σε βάθος. Εγώ έχω υποβάλει μια σειρά από τροπολογίες για το ζήτημα αυτό και θα ήθελα να ζητήσω από τις εισηγήτριες και από τις σκιώδεις εισηγήτριες όλα αυτά να τα εξετάσουν. Εγώ είμαι νομικός και δεν μπορώ να αγνώ όλες αυτές τις πτυχές του θέματος, τις προσπάθειες που κάνουμε. Ξέρετε πως υπάρχουν αυτά στις συνθήκες και πάνω στις συνθήκες θα πρέπει να βασίσουμε οποιαδήποτε ε, προσπάθεια κάνουμε. Άρα λοιπόν πλήρης ε, συμμόρφωση με τα όσα έχουμε στον κανονισμό Ρώμη 1. Και ένα τελευταίο σημείο Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει με τις τροπολογίες στον κανονισμό. Έχω κάθε διάθεση να προσπαθήσω. Αλλά για την επιβολή της τρέχουσας νομοθεσίας στα κράτη-μέλη, ρωτήστε με, ε, απαντήστε μου μάλλον, ποιος ασχολείται με το θέμα αυτό. Για τη Γαλλία, για παράδειγμα. Εκεί έχουμε ένα πρόσφατο διάταγμα, το οποίο εγκρίθηκε, το οποίο απαιτεί ε, να έχει κανείς ε, καλό επίπεδο γαλλικής γλώσσας για να μπορεί να δουλέψει κανείς στην οικοδομή. Και δεν μπορεί κανείς στον κατασκευαστικό κλάδο της Γαλλίας να δουλέψει εάν δεν μιλάει γαλλικά. Νομίζω ότι τέτοιου είδος φαινόμενο θα πρέπει να τα ε, πατάξουμε και εκεί ίσως είναι και η βασική μάχη που πρέπει να δώσουμε. Τώρα, θα ήθελα να κλείσω εστιάζοντας στο επόμενο σημείο γιατί πρέπει να σας πω ότι εδώ δεν μπορώ να ευθυγραμμιστώ με τα όσα προτείνουν οι συνεισηγήτριες. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε προσπάθειες να συμβιβαστούμε για την νομοθεσία αυτή είναι απαραίτητη. Κύριος Λέναρτς και μετά ο κύριος Κούγκαν. Κύριε Λέναρτς, σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τους, ε, τις συνεισηγήτριες για την ε, πολύ σκληρή δουλειά και για τους ε, ε συναδέλφους που υπέβαλαν 500 τροπολογίες. Θα ήθελα για μία ακόμα φορά, γιατί το έχω ξαναπεί, να πούμε ότι εδώ γίνεται λόγος για ελεύθερη κυκλοφορία και δικαίωμα εγκατάστασης. Δεν μιλάμε εδώ για δικαίωμα ελεύθερης εργασίας είναι ελεύθερη, υπηρεσία, ελεύθερη ε, μετακίνηση και παροχή υπηρεσιών. Ε, είναι γεγονός ότι εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερους ε, αποσπασμένους εργαζόμενους στην Ευρώπη και όχι λιγότερους. Και εγώ είμαι σε μεθόρια περιοχή και πραγματικά σας το λέω και σας το υπογράφω. Όμως χρειαζόμαστε καλύτερες συνθήκες για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Έτσι, ε, ε, ξέρετε, είναι δύο οι ομάδες. Είναι αυτοί που θέλουν να κάνουν την απόσπαση πιο εύκολη και αυτοί που θέλουν να κάνουν την απόσπαση πιο δίκαιη. Και επομένως θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ των δύο και αυτό ε, σας ε, συστήνω ε, τις δικές μου τροπολογίες γιατί πιστεύω ότι έχουν βρει τη χρυσή τομή. Να τις διαβάσετε λοιπόν με προσοχή. Κοιτάξτε, η απόσπαση εργαζομένων ε, δεν είναι ίδια με αυτήν που πιστεύαμε τη δεκαετία του 90 ε, γιατί οι συνθήκες έχουν αλλάξει και οι προϋποθέσεις είναι διαφορετικές. Ε, θα πρέπει λοιπόν πρώτον να ξεκαθαρίσουμε ποια δουλειά, ποια ανάγκη καλύπτει ο συγκεκριμένος αποσπασμένος οργάνος. Θα πρέπει να μιλήσουμε για την αμοιβή, λοιπόν δεύτερο θέμα και συμφωνώ απολύτως με τις προσπάθειες που καταβάλουν οι συγγήτριες έτσι ώστε ε, να ευθυγραμμιστούν οι διαδικασίες αυτές με τις εθνικές διαδικασίες και νομίζω ότι αν καταφέρουμε να ε, βρούμε ένα σωστό τρόπο να ορίσουμε την, αμυγή, ε, την αμοιβή σε αυτήν την οδηγία, τότε ταυτόχρονα θα λυθούν και πολλά θέματα. Αλλά όταν μιλάμε για τη διάρκεια τώρα, ε, νομίζω ότι και εκεί θα λυθεί το θέμα εάν το ζήτημα της αμοιβή είναι σαφές. Τέλος θα πρέπει να υπάρξει, να υπάρξει κάποια ευελιξία ανατομέα με την έννοια δηλαδή ότι όλοι οι τομείς δεν είναι οι ίδιοι. Υπάρχουν άλλοι που έχουν λιγότερη ανάγκη από τους αποσπασμένους, άλλοι που απασχολούν περισσότερους κτλ. Τελευταίο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι συμφωνώ απολύτως με τον προηγούμενο συνάδελφο. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι ε, γιατί αυτό που κάνουμε εδώ είναι ε, να ε, αποφασίσουμε για μία νομοθέτηση και για μία νομική βάση η οποία να είναι αυτάρκηση. Δηλαδή να μην ξεκινήσουμε με ένα νομοθέτημα το οποίο μετά θα χρειαστεί να γεννήσει άλλο. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κούκαν και μετά ο κύριος Μάν. Κύριε Κούκαν παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ ιδιαίτερος και συγχαρητήρια στις δύο εισηγήτριε για την πολύ καλή δουλειά και τη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε σήμερα, αλλά ταυτόχρονα και για όλους και προς όλους ε, για τις προσπάθειές τους ένα πολύ δύσκολο και πετητικό θέμα. Κάποιες πιο γενικές παρατηρήσεις. Τις ε, μου, τις ειδικότερες, τις εκφράζουμε από τις τροπολογίες μου, άλλωστε. Πρέπει το θέμα της μεταφοράς, των μεταφορών να καλύπτεται από ειδικέ τομεακές αποφάσεις και καλό τις εισηγήτριες να αναλογιστούν τι είδους συνέπειες θα έχει αυτό για τις επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση δεν πρέπει να είναι ε, μια αντιπαράθεση μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Έχει περισσότερο σαν στόχο να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της ενιαίας αγοράς αμφίδρομα. Πάνω απ' όλα όμως να διαφυλάξει την ελευθερία κυκλοφορίας και παροχής υπηρεσιών. Πρέπει λοιπόν για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος να αφουγκραστούμε περισσότερο αυτούς οι οποίοι έχουν ε, την καθημερινή εμπειρία από τις αποσπάσεις και βέβαια τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που αποσπούν εργαζομένους αλλά και τους αποσπωμένους εργαζομένους και πάνω απ' όλα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να μην επιβληθεί επιπλέον φόρτος γραφειοκρατικός ούτε για τους μεν ούτε για τους δε. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Mann. The floor is yours. And uh, after you it... Ο κύριος Μαν και μετά η κυρία Γιώσουβικ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συνεισηγήτριες ε, θερμά βλέπουμε από όλες τις τοποθετήσεις ότι είναι σαφής η πρόθεση για εξασφάλιση συμβαστικής λύσης που θα ικανοποιεί και τις μεγαλύτερες αλλά και τις μικρότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακούστηκαν κάποιες γενικές αρχές. Πάνω από όλα δεν πρέπει να επιτρέψουμε πουθενά το κοινωνικό τάμπινγκ. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να καταστεί απόλυτο σαφές μέσα σε αυτή την οδηγία αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να επιτρέψουμε ούτε και τον προστατευτισμό που βλέπουμε να αναδύεται και πάλι από τις Ηνωμένε Πολιτείες και από τη νέα ηγεσία τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποτρέψουμε να μεταδοθεί στην Ευρώπη. Η απόσπαση πρέπει να είναι γνήσια και όχι πλασματική. Και αυτό θα κριθεί από το διάστημα που θα περνά στη χώρα υποδοχής ο αποσπασμένος εργαζόμενος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τις καταστρατηγήσεις, δεν πρέπει να επιτρέψουμε τις εταιρείε γραμματοθυρίδα, γιατί αυτό δεν είναι αμεληταίο ζήτημα, είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν μπορούμε καν να ισχυριζόμαστε ότι πια δεν γνωρίζουμε τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό και μην ξεχνάμε το θέμα των εγγράφων του Καναδά. Έχω ε, συμμετάσχει στη σχετική επιτροπή και έχει άμεση συνάφεια το θέμα των εταιριών γραμματοθυρίδων. Γιατί, γιατί επιτρέπουν σε ορισμένους να αποκρύπτουν ε, δραστηριότητες και έσοδα, ενώ οι μικροί μεσαίοι, οι οποίοι τηρούν τους κανόνες, βρίσκονται πάντα σε πιο μειονεκτική θέση. Πρέπει λοιπόν να είναι σαφές το ποιος είναι ο εταίρος και βέβαια και ποιος είναι και ο ε, κοινωνικός εταίρος, αν προκειμένου. Κάτι το οποίο δεν έχω ακριβώς αντιληφθεί από κάποιες από τις ε, τροπολογίες που είδα ήταν αντιπροσωπευτικές η λέξη συλλογικές συμβάσεις. Τι σημαίνει αντιπροσωπευτική συλλογική σύμβαση, δηλαδή αντικαθιστά τη συλλογική σύμβαση, πώς κρίνεται αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Λοβιέκα. Και μετά Βέμπερ. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους για τις τροπολογίες, η ευρεία πλειονότητα των οποίων αποδεικνύει πως όλοι επιδιώκουμε σαφείς και διαφανείς διατάξεις για την απόσπαση των εργαζομένων ώστε να προχωρήσει κατά τρόπο ασφαλή η νομοθεσία στην Ευρώπη. Κοιτάω λοιπόν τις ε, τροπολογίες από πλευράς της ομάδας μου προσπαθώ να συντάξω κείμενα τα οποία θα είναι σαφή και κατανοητά και απλά για τους εργαζομένους αλλά και τους εργοδότες. Προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τις νομικές συνέπειες οι οποίες θα ακολουθήσουν τη μεταβατική περίοδο των 24 μηνών. Προτείνουμε νέα δικαιώματα που θα μπορούσαν να ε, αναγνωριστούν στον αποσπασμένο εργαζόμενο, άρθρο 29, μεγαλύτερη ευελιξία στον υπολογισμό της ε, περίοδου απόσπασης αντί για 24-36 μήνες και δυνατότητα και για παρεκκλήσεις και δυνατότητα διακοπής για δύο μήνες στην περίοδο αυτή, όπως άλλωστε προβλέπει η νομοθεσία κάποιων από τα κράτη. Ε, προτείνουμε επίσης ε, ρήτρα ε, καλύτερου που θα επιτρέψει μάλλον καλύτερο συντονισμό με τον κανονισμό 823 και όταν καλύπτεται ένας αποσπασμένος εργαζόμενος από την κοινωνική ασφάλιση της χώρας στην οποία εργάζεται, στην οποία είναι αποσπασμένος, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτή η διάσταση. Στην τροπολογία 365 επίσης σημειώνουμε ότι θα πρέπει πέραν των ελάχιστων αμοιβών να υπάρχει αποζημίωση για ε, ε, παραμονή στην, ε, στο χώρο της, στον τόπο της απόσπασης του εργαζομένου σε περιόδους επίσημων αργιών και τα λοιπά. Και βεβαίως τα πρόσθετα αυτά στοιχεία θα πρέπει να τα προσδιορίσουν τα κράτη-μέλη. Η 412 επίσης είναι πολύ σημαντική τροπολογία. Αφορά την υποχρέωση δημοσίευσης των πληροφοριών σε ιστότοπο για να μπορεί να κάνει τον υπολογισμό πέραν του ελάχιστου μισθού της ελάχιστης αμοιβής ο και των πρόσθετων που μπορεί να περιμένει. Οι μεταφορές πρέπει να αποκλειστούν. Μιλούμε για ναυσιπλοεία μικρών αποστάσεων και διαμετακόμιση. τομείς ειδικού δηλαδή και υπηρεσίες που θα πρέπει να καλυφθούν από τομεακούς κανονισμούς. Επανελειμμένος μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σημειώσει ότι δεν θα πρέπει το θέμα αυτό να ενταχθεί και οι μεταφορές αυτές να θεωρηθούν ε, ε, ισότιμες με οποιοδήποτε άλλο είδος απόσπασης. Επίσης σημειώνουμε, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ότι η συντριπτική πλειονότητα των αποσπάσεων έχει να κάνει με προέλευση και απόσπαση σε δυτικά κράτη. Ευχαριστώ πολύ, Βέμπερ και μετά Σόιντροβα. Θα ήθελα να πω πως εκτιμώ ιδιαίτερα τη σκληρή δουλειά που έχουν κάνει όλοι οι συνάδελφοι για το συγκεκριμένο θέμα ανεξάρτητα με το ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις για κάποια θέματα. Και θα ήθελα να σας πω το εξή. Για μένα υπάρχει ένας βαθμός σύγχυσης. για το για ποιο λόγο έχουμε προχωρήσει σε αναθεώρηση αυτής της οδηγίας και τελικά ίσως καταλήξουμε σε μια διαίρεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα ωφελήσει κανέναν. Καταρχήν αν εξετάσει κανείς τα ταστιστικά δεδομένα θα δει πως οι αποσπάσεις είναι κυρίως θέμα δυτικών με δυτικές χώρες ενώ με στη Δυτική Ευρώπη. Αυτοί όμως οι οποίοι επηρεάζονται ως ε, ε, παράπλευρες απώλειες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις ε, χωρίς κεντρικής Ευρώπης. Γιατί όλες αυτές οι απαιτήσει, οι σκληρές προϋποθέσεις σημαίνουν ότι μόνο οι, οι πολυεθνικές και οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορέσουν στις αγορές αυτές να επιβιώσουν. Ένα ακόμα σημείο σύγχυσης. Το γεγονός πως έχουμε συγχύσει την... Ε, ότι συγχαίρουμε την ιδέα της προστασίας του εργαζομένου που είναι ε, πολύ σωστό, με ε, την ε, τιμωρία παράνομων πράξεων. Μα αν είναι παράνομη μια πράξη υπάρχουν κυρώσει. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να μιλάμε για παράνομες πράξεις και μετά να φέρνουμε νομοθεσία για την απόσπαση εργοζομένων. Τι σχέση έχει μια παράνομη με μια νόμιμη ενέργεια και για τον Πολωνό υδραυλικό. Μα δεν έχει πάρει ποτέ απόσπαση ο καημένο. Είναι ένα εργαζόμενο υδραυλικό που αποφάσισε να φύγει από τη χώρα του και να πάει αλλού όπω οποιοδήποτε άλλο εργαζόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά τα αναφέρουμε μέσα στην ε, οδηγία περί απόσπασης προσπαθώντας να λύσουμε προβλήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να ακουμπήσουμε κατά τη γνώμη μου. Και αυτό μας οδηγεί στη νομική βάση. Γιατί στην απόσπαση εργαζομένων η νομική βάση σχετίζεται με την υπηρεσία. Και νομίζω ότι υπάρχουν διάφοροι μύθοι που μας οδηγούν στη διεύρυνση της νομικής βάσης και γι' αυτό ε, προτείνω ε, να μην ε, προχωρήσουμε και να αλλάξουμε τη νομική βάση. Επίσης θεωρώ πως Χρειαζόμαστε ε, για τις μεταφορές συγκεκριμένη νομοθεσία, αλλά για τις μεταφορές να σας πω πως ήδη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την κεντρική Ευρώπη έχουν χάσει την ευρωπαϊκή αγορά. Δεν μπορούν πλέον να προσφέρουν ε, Υπηρεσίε γιατί δεν μπορούν πια να γνωρίζουν νομοθεσία σε όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί δεν είναι μόνο οι νόμοι, είναι και τα, το διοικητικό δίκαιο και το περιφερειακό και το τοπικό δίκαιο που δεν το βλέπετε ποτέ σε καμία ιστοσελίδα και στο τοπο, ε, τοπικής ε, διοίκησης. Και έχω μιλήσει με πάρα πολλέ ενώσει ε, μεταφορικών εταιριών, συνδικάτων κτλ. Και πρέπει να σας πω πως έχουμε περιπλέξει τη ζωή τους σε μεγάλο βαθμό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σόιντροβα και μετά κυρία Στίβενς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια συζήτηση που δίνει μια ευκαιρία να εξηγήσουμε τις τροπολογίες μας. Αν θέλουμε η οδηγία να είναι διάφανη, θα πρέπει εμείς να μπορούμε να εξηγήσουμε το σκεπτικό μας και γιατί προτείνουμε όσα προτείνουμε. Εγώ κατέθεσα 11 τροπολογίε και θα εξηγήσω μόνο δύο από αυτέ. Πρώτα απ' όλα, για την νομική βάση πιστεύω πως η νομική βάση θα πρέπει να διευρυνθεί για να καλύψει και την προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων αλλά να υπογραμμίσουμε πως υπάρχει νομική βάση η οποία είναι η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών. Άρθρο 56 να επιστρέψει παρακαλώ στο κείμενο και να αναφερόμαστε ρητά στην ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών. Και η δεύτερη τροπολογία είναι αυτό του κλάδου των μεταφορών. Ο συμβιβασμός λοιπόν όλων των διαφορετικών τροπολογιών που σχετίζονται με τη μεταφορά είναι μια πρόταση μέσω της οποίας προσπαθώ να εξηγήσω πως η οδηγία του 96 θα πρέπει να ισχύει μέχρι τις προτάσεις της Κομισιόν για νέα νομοθεσία που θα είναι ε, συγκεκριμένη για συγκεκριμένο κλάδο, δηλαδή στην περίπτωση αυτή τον κλάδο των μεταφορών. Να το πω διαφορετικά. Δηλαδή, το διοικητικό βάρος που αυξάνεται και το οποίο ε, η αναθεώρηση αυτή εισάγει δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί στον κλάδο των μεταφορών και όλοι κατανοούμε και οι συγητές μας επιβεβαιώνουν πως οι μεταφορές είναι ένας πολύ συγκεκριμένο κλάδος που χρειάζεται τη δική του νομοθεσία. Άρα λοιπόν η αναθεώρηση αυτής της οδηγίας δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται για τις μεταφορές. Οι μεταφορές θα πρέπει να μείνουν υπό την εντολή της οδηγίας του 96. Thank you. Ε, the floor to Madam Helga Ευχαριστώ πολύ κυρία Helga Stevens και μετά τελευταίος ο μιλητής. Ε, ο κύριος Κρίστινσέν. Κυρία Στίβενς, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη γιατί μπερδεύτηκα προηγουμένω. Ε, εγώ σκεφτόμουν να ε, αναφερόμουν σε ένα άλλο ε, θέμα για το οποίο είμαι σκιώδη, αλλά που θα το μελετήσουμε το απόγευμα. Εν πάση περιπτώσει, ζητώ συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω τι δύο εισηγητρίε για την εργασία που έκανα σε, αυτή την εξαιρετικά αυτό το εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Επίση, να πω ότι είναι απολύτω απαραίτητο ε, να συνεχίσουμε την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ. Αυτό είναι πραγματικά θεμελιώδου σημασία για την προστασία των εργαζομένων. Ε, επίσης, ε, να μην λησμονούμε ότι είναι σημαντικό και για την εικόνα που δίνουν οι πολίτες, που έχουν συγγνώμη, οι πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους πολίτες. Έχω κάποιες ε, παρατηρήσεις ε, εξορισμού η μετακίνηση αυτού του είδους ε, είναι συγκεκριμένη, έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και πιστεύω λοιπόν ότι για να αποφύγουμε και το κοινωνικό ντάμπινγκ θα πρέπει να επιβάλλουμε τη μέγιστη δυνατή διάρκεια η μέση διάρκεια μιας απόσπασης είναι λιγότερη από τέσσερις μήνες και επομένω θεωρώ ότι μια καλή πρόταση είναι το εξάμεινο. Ε, τώρα, το ποιο τομέα είναι τομέα κινδύνου πρέπει να αποφασιστεί από τα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, η προσέγγιση αυτή ε, σέβεται την αρχή της επικουρικότητας. Κατά την άλλη πλευρά, κατά, <laughs> την άλλη πλευρά ε, είναι γεγονός ότι μέσω της ε, ε, απόσπασης πολλές χώρες έχουν βελτιώσει την οικονομική τους κατάσταση. Δεν ταυτίζεται απαραίτητα η απόσπαση με το κοινωνικό ντάμπινγκ. Γι' αυτό λοιπόν δεν πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να καλύψουμε, να εφαρμόσουμε μάλλον και να επιβάλλουμε μέγιστη διάρκεια σε τομείς που δεν αποτελούν τομείς κινδύνου. Βεβαίως θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την κοινωνική απάτη, αλλά δεν θα πρέπει ε, να ακυρώσουμε τα καλά της ε, ελευθερίας κίνησης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε ξανά το θέμα αυτό και σε συνάρτηση και με τη μεταρρύθμιση της οδηγίας για την κοινωνική ασφάλιση. Επίσης, η αρχή της ίση αμοιβή ε, για ίδια εργασία στον ίδιο τόπο εργασία. Αυτό είναι από τον Ουκάνεφ και θα είναι ένα σημαντικό βήμα προ την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ και της κοινωνική απάτης. Ε, ε, Αδιαφυσβήτητα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δημιουργήσει θέσει εργασία και ευημερία και όχι να αποτελέσει την αιτία καταστροφή και απώλειας θέσεων εργασία ούτε να προκαλέσει την καταστροφή κάποιων χωρών. Απ' την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε και οι κανόνες που διέπουν την ε, αμοιβή ε, πρέπει να είναι απλοί και ε, διάφανοι. Επίσης, εάν οι κανόνες είναι ιδιαίτερα περίπλοκοι και αν το διοικητικό και λοιπόν είναι ιδιαίτερα βαρύ, τότε δύσκολα θα εφαρμοστούν καλά. Εγώ πιστεύω ότι με σωστή εφαρμογή τη οδηγία για του ε, αποσπασμένου εργαζόμενου θα έχουμε αποτελεσματικότερη ενιαία αγορά. Και επαναλαμβάνω ότι το, υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να παραμείνουν εθνική αρμοδιότητα. Όπω και ο προηγούμενο ομιλητή είπε, θα πρέπει να, δημιουργήσουν, να δημιουργήσουμε καλέ συνθήκε και ευκαιρίε για όλου. Ε, και εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω αυτήν την διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Στίβενς. Κύριε αν έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ βεβαίως τις εισηγήτριες για την εξαιρετική δουλειά. Η βάση εκκίνησης είναι πολύ καλή, την κατανομή σε δύο τίτλους. Μπορούμε να εντοπίσουμε καλύτερα κάποιες δυσκολίες που αφορούν την οδηγία. Βεβαίως, όπως είπε και ο κύριος Μαν, πρέπει και τον προστατευτισμό να καταπολεμήσουμε και, την, και το κοινωνικό ντάμπινγκ. Αυτό μπορεί συνθήκη δηλαδή. Ισότιμη μεταχείριση, χωρίς διακρίσεις. Και αυτή θα πρέπει να είναι και η κόκκινη γραμμή. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να καταστρατηγούνται αυτοί οι κανόνες και δεν θα συμφωνήσω με εκείνους που λένε ότι ε, θα πρέπει να αποκλειστούν οι μεταφορές από το πεδίο εφαρμογή. Βεβαίω θα υπάρξει κάποια εξειδίκευση ως προς τον τομέα των μεταφορών, αλλά το εργατικό δυναμικό που αποσπάται και στο χώρο των μεταφορών θα πρέπει να καλύπτεται από την Γενική Οδηγία. Δεν μπορεί να ισχύει τίποτε άλλο. Άλλωστε αυτό πιστεύω αποτελεί και μια καλή δοκιμασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδικότερα, θα κριθεί από το αν μπορούμε να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων και να εξασφαλίσουμε μια καλή πλειοψηφία υπέρ της οδηγίας χωρίς σοβαρού ε, σοβαρούς διχασμούς εσωτερικούς. Το ίδιο θα είναι δοκιμασία βέβαια και για το Συμβούλιο των Υπουργών. Να δούμε αν θα μπορέσουν χωρίς να διχαστούν μεταξύ τους τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν ένα κείμενο οδηγίας. Γιατί ναι, είναι πολλές βέβαια οι διαφορές μέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά όχι τόσο βαθιές. Ενώ στο Συμβούλιο φαίνεται ότι είναι τέτοιες οι διαφορές που ίσως να μπορέσει να προκύψει καν αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, που ήσασταν και τόσο σύντομος και σαφής. Μπορούμε να δώσουμε λίγα λεπτά την Επιτροπή και θα σας αφήσουμε, θα σας αφήσουμε εσάς τα υπόλοιπα 25 λίγο πολύ. Κύριος Περέιρα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Καταρχάς ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε. Ευχαριστούμε τις δύο συνεισηγήτριες. Εξαιρετική δουλειά τους. Και βεβαίως ευχαριστώ όλους τους βουλευτές για τις προσπάθειές τους ε, για τη σύνταξη τόσων τροπολογιών. Πάλι θα μείνω και εγώ στο σχόλιο της κυρίας Μωρέν Σαχτιέ ότι είναι μικρές οι αποκλήσεις σε σχέση με τον όγκο και τη σοβαρότητα του θέματος. Δεν θα τοποθετηθώ στις τροπολογίες, άλλωστε δεν είναι αυτός ο ρόλος μου, αλλά θα μου επιτρέψετε να κάνω κάποιες γενικές ε, παρατηρήσεις που είναι σημαντικές ως προς την αντίληψη που θα έχουμε των τροπολογιών. Καταρχάς, συμφωνούμε απολύτως με αυτό που υπογράμμισαν οι δύο συνεισηγήτριες και πολλοί βουλευτές, ότι χρειάζονται σαφείς κανόνες. Κανόνες που θα μπορούν να ελέγχονται κατά την εφαρμογή τους. Αυτό και εν παρόδο υπογραμμίζω ότι η πρόταση που κάνουμε για τις αμοιβέ αυτό το στόχο επιδιώκει όντας βέβαια ταυτόχρονα και διατεθειμένοι να υπογραμμίσουμε ότι τροπολογίες που έχουν ε, σαν στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας για τις συνθήκες εργασίας που εφαρμόζονται, που ισχύουν για τους αποσπασμένους εργαζομένους υπό την ε, νέα οδηγία, επίσης θα διευκολύνουν την συγκεκριμένη εφαρμογή της νομοθεσίας και άρα βαίνουν προς την ορθή κατεύθυνση. αντίον, η διάχυση διαφόρων, ο πολλαπλασιασμός διαφορετικών συστημάτων που θα ισχύουν για τους εργαζομένους αναλόγως ε, διαφορετικών χρονικών περιόδων κτλ. Ε, μάλλον τίνουν προς την εσφαλμένη κατεύθυνση. Εάν έχουμε δηλαδή άλλο πακέτο κανόνων που ισχύουν για όποιον εργάζεται μέχρι έξι μήνες, άλλο για εκείνον που εργάζεται περισσότερο ή λιγότερο κτλ. Δεν εξυπηρετούμε ούτε τις επιχειρήσεις, ούτε τους εργαζομένους, ούτε και τις επιθεωρήσεις εργασία. Και επίσης είναι σημαντικό πιστεύω να διαφυλαχθεί ο αρχικός στόχος της οδηγίας που είναι ο συντονισμός των εθνικών νομοθεσιών που ορίζουν τις συνθήκες τις ε, ισχύουσες για τους αποσπασμένους εργαζομένους για να λειτουργήσει καλύτερα η παροχή των υπηρεσιών αυτών και η ενιαία αγορά βεβαίως και ο συντονισμός θα πρέπει να γίνεται αυστηρά κατά την περίοδο της απόσπασης. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτό το όριο, ότι δηλαδή η οδηγία ε, ορίζει συζητά, αντιμετωπίζει συνθήκε εργασία και μόνο για την περίοδο τη απόσπαση. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιε προσπάθειες μέσα από τι τροπολογίε να επιβληθούν ρυθμίσει σε τομεί ε, ή θέματα που δεν αφορούν αυστηρά την περίοδο τη απόσπαση και μπορεί να αφορούν την περίοδο που προηγείται τη απόσπαση ή μια άλλη χρονική περίοδο που μπορεί να ακολουθεί ενδεχομένω την απόσπαση. Λοιπόν, είναι μεγάλος επιδεσμό, το καταλαβαίνουμε, αλλά πρέπει να αντισταθούμε σε αυτόν και ε, να αφορά η νέα νομοθεσία αυτή, η οδηγία αυτή αυστηρά και μόνο την περίοδο της απόσπασης. Αυτός όλος είναι ο στόχος της οδηγίας. Επίσης, έχω τονίσει και στο παρελθόν, θα το επαναλάβω, γιατί είναι πολύ σημαντικό ε, και εν ώψη της νομικής βάσης και εν ώψη του στόχου της οδηγίας, ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε την εισαγωγή κανενός κανόνα που με κάποιο τρόπο θα επέβαλε διαφορές μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών ε, ε, σε εσωτερικό εθνικό επίπεδο και εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες πέραν των συνόρων. Ε, αυτό είναι το νόημα κάποιων τροπολογιών όπως τις διαβάζω. πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερος ώστε οι συνθήκες εργασίας που γίνονται δεκτές για τους αποσπασμένους εργαζομένους να μην στηρίζονται σε διατάξεις τόσο ευρείες που τελικά να είναι πιο αυστηρές συνθήκες για εκείνους που παρέχουν πέραν των συνόρων υπηρεσίες ε, σε σχέση με αυτούς που μένουν στα εθνικά σύνορα. Αυτό και μια τελευταία παρατήρηση για να υπενθυμίσω. Ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό νομικά τη νομική βάση. Μπορεί βέβαια να έχει και την πολιτική τη σημασία, αλλά υπάρχει ευρύτατη νομολογία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα κριτήρια πάνω στα οποία θα κριθεί, θα ε, ε, επιλεγεί η νομική βάση. Και βέβαια σε αυτά τα κριτήρια είναι και η ε, συνέχεια του νομοθετήματος. Επίσης η νομολογία τονίζει παγίως ότι διπλές νομικές βάσεις μόνο κατά εξαίρεση μπορούν να επιβάλλονται, μόνο όταν δηλαδή υπάρχει, υπάρχουν δύο τελείως ασυμβίβαστες νομικές βάσεις που μόνο σε συμπληρωματικό ρόλο μπορούν να υπάρξουν ή απαιτείται να υπάρξουν. Υπογραμμίζω για άλλη μια φορά ότι στόχος της οδηγίας είναι να επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία της, ενιαία, της ιστορικής αγοράς, συντονίζοντας τις εθνικές νομοθεσίες για τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων. Αυτή είναι η βάση. Και νομίζω ότι αυτό το έχει ήδη εντοπίσει η νομολογία του δικαστηρίου και το κυρίαρχο στοιχείο ακριβώς που θα ορίσει την νομική βάση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιονγκέριος και κυρία Μογαν Έχουν στη διάθεσή τους ακόμα 23 λεπτά για τα συμπεράσματα. Κυρία Ιονγκέριος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έδωσαν αυτή την επιπλέον διάσταση σε κάτι έτσι κι αλλιώς θα είχαμε διαβάσει γραπτά. Άρα λοιπόν χαίρομαι ιδιαίτερα που όχι μόνο διαθέσατε το χρόνο να διατυπώσετε αυτές τις τροπολογίες, αλλά να μας παρουσιάσετε εδώ αυτό το επιπλέον χρώμα ε, και να εξηγήσετε ακριβώς τι εννοείτε με τις τροπολογίες σας. Ελπίζω πως στο άμεσο μέλλον δεν θα τρομάξετε όταν σας ζητήσω για μια φορά ακόμα να μας εξηγήσετε το υπόβαθρο στο οποίο βασίζονται σε αυτές τις τροπολογίες, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, Όντως, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Όμως, αισθάνομαι βέβαιη πως θα τα καταφέρουμε όλα. Και αυτό θα γίνει βέβαια ε, πώς, ακούγοντας τις δικές σας προτάσεις και προσπαθώντας να βρούμε αυτή τη χρυσή τομή, τον κοινό τόπο που θα μας επιτρέψει στο μέλλον να προχωρήσουμε έτσι ώστε να έχουμε μια καλή, ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς που θα συνδυάζεται με τη σωστή μεταχείριση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά παράλληλα και με την ορθή μεταχείριση των εργαζομένων. Αυτό δηλαδή απαιτεί μια λεπτή ισορροπία, την οποία εμείς θα πρέπει να επιδιώξουμε και βέβαια αυτό το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να καταθέσουμε τα όπλα, να πούμε πως εμείς δεν θα τα καταφέρουμε Γιατί ξέρετε, να το πω έτσι, οι πολίτες μας πληρώνουν μια πολύ γερή αμοιβή για να μπορούμε να το καταφέρουμε, για να μπορούμε να βρούμε λύσεις. Νομίζω λοιπόν ότι για όλους μας και για εμένα σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια την ελευθερία της κυκλοφορίας των εργαζομένων που αποτελεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων. Δεν θέλουμε αυτό για οποιοδήποτε λόγο να πάψει να ισχύει. Και νομίζω πως εγώ στο παρελθόν, επειδή ήμουν ε, συνδικαλίστρια ε, σε ηγετική θέση, το να ε, θέλεις να μεταφερθείς κάπου αλλού για να δουλέψει, είναι θεμελιώδε δικαίωμα το οποίο θα πρέπει να μπορεί να ασκήσεις, να πας ε, κάπου αλλού, να βρει ευκαιρίες εργασιακή. αν πιστεύεις πως αυτό ε, θα σου προσφέρει κάτι. Υπερβολικά συχνά. Πια η ελευθερία, η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ε, ουσιαστικά καταπατάτε ή μάλλον γίνεται μια κακή χρήση αυτής, όχι έτσι ώστε να προστατεύσει τους εργαζόμενους, αλλά για να καταπατήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα αυτών. Νομίζω λοιπόν το πιο σημαντικό για μας είναι να βρούμε μία ισορροπία μέσω της κατάλληλης πρότασης. Δεν θα απαντήσω σε όλες τις προτάσεις ε, με συγκεκριμένη απάντηση, γιατί αυτό θα έδινε την εντύπωση ότι γνωρίζω πού θα βρούμε τη χρυσή τομή. Και βέβαια έχω και τη δική μου θέση, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό να εξετάσουμε πώς μπορούμε να βρούμε αυτό τον κοινό τόπο που θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε μια συνενετική θέση στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή πρώτα να ψηφίσουμε εμείς και χαίρομαι γιατί έχω την αίσθηση ότι και από το Συμβούλιο λαμβάνω κάποια θετικά μηνύματα. Αν λοιπόν το Συμβούλιο ακολουθεί το ίδιο χρονοδιάγραμμα με εμάς, τότε εφόσον τελειώσουν εκεί οι εργασίες θα μπορέσουμε να μπούμε στον τριμερή διάλογο και για να γίνει αυτό χρειάζεται ακριβώ να έχουμε μια ιδρία συνένεση εδώ. Νομίζω πως είμαστε υποχρεωμένοι να τα καταφέρουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε από τα αποτελέσματα, αποτελέσματα που αυτή τη στιγμή θα μας επιτρέψουν να αποφύγουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ, αλλά θα μας βοηθήσει όλους επίσης να αποφύγουμε οποιοδήποτε προστατευτισμό. Και θα κλείσω λέγοντας πως επιτρέψτε μου Όποτε θέλω να σας τηλεφωνήσω για να σας ζητήσω διευκρινήσεις για την ε, κατάσταση των τροπολογιών και με μεγάλη χαρά αναμένω όχι μόνο να συνεργαστώ με τη συνεισηγήτριά μου αλλά και με τους σκιώδεις και όσους βρίσκονται εδώ στην Επιτροπή μας. Επ' αυτής της μάλλον ε, ευρείας βάσης και βέβαια Θα το γράψω και πάνω από το γραφείο μου. Πρέπει να το καταφέρεις. Euh, Ευχαριστώ πάρα πολύ Αγνέσα για αυτή την πολύ ανοιχτή ε, και ε, αισιόδοξη τελευταία φράση. Και εγώ να πω δύο λόγια για να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, όλους τους συναδέλφους επίσης που μίλησαν σήμερα το πρωί, ε, έτσι ώστε να διαλευκάνουν, να διευκρινίσουν ακόμα περισσότερο μάλλον την ε, επιχειρηματολογία τους. Το πρώτο σημείο το οποίο με εκπλήσει είναι ότι ε, το συλλογικό πνεύμα αλλάζει. Αυτό το οποίο συγκρατώ ε, γιατί πραγματικά ακούγοντάς σας έκανα πολλές, πήρα πολλές σημειώσεις και σας λέω μερικές από τις φράσεις που είπατε. Δεν θέλουμε να χωρίσουμε την Ευρώπη. Αυτό το επικ οικοδομητικό ε, συνολικό ευρωπαϊκό πνεύμα νομίζω ότι ε, ήταν προφανές ε, από τις σημερινές παρεμβάσεις και είναι γεγονός ότι πρέπει να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα θετικό συμπέρασμα και για να φτάσουμε στο θετικό συμπέρασμα πρέπει γενικότερα η διάθεσή μας, η προσέγγισή μας να είναι θετική, να μην μοιράσουμε την Ευρώπη, να την ενώσουμε ακόμα περισσότερο. Άκουσα και επεξηγήσεις και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί πολλοί από εσά είδατε ότι η Γαλλία, η χώρα από την οποία προέρχομαι, την προηγούμενη εβδομάδα ε, έχει ανησυχήσει πάρα πολύ από τη λεγόμενη ρήτρα μολιέρου, δηλαδή τη ρήτρα που λέει ότι πρέπει να ξέρουν οι ξένοι εργαζόμενοι τα γαλλικά. Ε, και ε, ήθελαν κάποιοι, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, προσέξτε, γιατί στον, στο, στη Βουλή και στην ε, Γερουσία καταφέραμε να μπλοκάρουμε ε, αυτή τη ρήτρα η οποία ήταν πραγματικά ε, κατάφερη παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας, της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κτλ. Αλλά αλλά μπορεί να ληφθούν παρόμοιες αποφάσεις σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει να σας πω ότι αγωνίστηκα με νύχια και με δόντια κατά αυτής της λεγόμενης ρήτρα μολιέρου, ρήτρα ε, γαλλογνωσίας σε πάση περιπτώσει και ποτέ δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι κατά αυτής ή παρομοίων ρητρών. Γιατί έτσι αρχίζει και ε, ξυλώνεται σιγά σιγά η ελεύθερη κυκλοφορία, η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, ε, η ελευθερία εν τέλει των εργαζομένων. Ε, και πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει να έχετε ούτε μια στιγμή την παραμικρή αμφιβολία ότι εγώ θα υψώσω το ανάστημά μου πάντα απέναντι σε τέτοια πράγματα. Εγώ προσωπικά και το κόμμα μου αντιταχτήκαμε. Αλλά ξέρετε, είναι μία μάχη την οποία δεν θέλω να ξαναζήσουν άλλοι συνάδελφοι στις χώρες τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιο είναι το πνεύμα εργασίας που έχω εγώ, που έχουμε εμείς οι δύο. Ε, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή την, ε, το αφήγημα ε, Δύση εναντίον Ανατολή, Ανατολή εναντίον Δύση. Έχουμε μονάχα την Ευρώπη. Επομένω αυτή η ρήτρα ε, τη ε, γνώση τη γαλλική γλώσσα ευχαριστώ δεν θα πάρω. Και ε, νομίζω ότι πρέπει να σας πω για μία ακόμα φορά ότι η δέσμευσή μου, η στράτευσή μου είναι πλήρης και αταλάντευτη. Γιατί αντιτάχτηκα εγώ προσωπικά σε αυτή τη ρήτρα, αλλά στην ουσία ε, προστατεύω και εσάς και όλους τους εργαζόμενους που θέλουν να κινηθούν στην Ευρώπη. Δεύτερο, και χαίρομαι που λέω ότι και εγώ και η Ανιές αισθανθήκαμε το ίδιο πράγμα, δηλαδή ότι και εσείς όπως και εμείς προσπαθείτε να βρείτε τα σημεία συνένεσης. Δεν θέλουμε προστατευτισμό, θέλουμε να οικοδομήσουμε όμως μία συνένεση. Και άλλωστε το είπε και ο Σράφος Κρίστενσεν στην προσπάθεια εξέβρασης αυτής της συνένεσης θα είναι τελικά να βρούμε τη θέση του, του Κοινοβουλίου απέναντι στη θέση του Συμβουλίου. Ε, θέλουμε την ε, πλειοψηφία και θέλουμε ικανή πλειοψηφία έτσι ώστε να είναι ισχυρή η φωνή μας στον τριμερή διάλογο και αυτό θα πρέπει να γίνει αν θέλετε όπως και εμείς να κερδίσουμε ε, σε αυτό το θέμα. Δουλέψαμε πολύ μέχρι τώρα αλλά πολλά ακόμα πρέπει να κάνουμε. Όλοι μας, όχι εμείς οι δύο συνεισηγήτριες, όλοι μας πολλά έχουμε να κάνουμε. Και γι' αυτό απαντώ στην ε, Μαρτίνα που είπε ότι δεν συναντήθηκαν οι ε, σκιώδεις και να της πω ότι στην επόμενη, ε, ότι περιμέναμε πριν ορίσουμε την επόμενη συνεδρίαση των σκιωδών να έχουμε και όλες τις ε, τροπολογίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε ποιες δυνατότητες συμβιβαστικών λύσεων και τροπολογιών υπάρχουν. Και ε, ε, ενδεχομένως θα λάβετε μία πρόσκληση, ίσως εστάλει και χτες, δεν ξέρω, περιμένω επιβεβαίωση και από τη γραμματεία, ε, για σύγκληση συνεδρίαση συντονιστών την 5η Απριλίου. Τώρα ξεκινάει λοιπόν μια νέα φάση εργασίας, η αντιμετώπιση λοιπόν των τροπολογιών, η προσπάθεια οικοδόμησης συνένεσης, να δούμε πού μπορούμε να βρούμε τα συνενετικά σημεία Είμαστε ανοιχτοί ε, και βεβαίως δεν υπάρχει μία συνένεση χοντροκομμένη, υπάρχουν σημεία επί των οποίων μπορούν να δημιουργηθούν, να οικοδομηθούν διαφορετικές πλειοψηφίες. Αυτό που εγώ θεωρώ σημαντικό είναι να συζητήσουμε ε, και να αντιμετωπίσουμε μεταξύ μας την εγγύηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ως πολιτική γραμμή να έχουμε οπωσδήποτε την αρχή ίση αμοιβή για ίδια εργασία, γιατί διαφορετικά οπωσδήποτε θα οδηγηθούμε σε πλήρη καταστρατήγηση των κοινωνικών αρχών, ε, να βρούμε μια λύση όσον αφορά το θέμα της αμοιβή. Οπωσδήποτε επίσης θα έχουμε ε, τέτοιες συζητήσεις όσον αφορά τη διεύρυνση της νομικής βάσης. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την πρόνοια του κυρίου Περέιρα, του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας είπε ότι οι ε, διπλές νομικές βάσεις ε, ε, αποφασίζονται μόνο και αποκλειστικά κατ' εξαίρεση. Έχετε δίκιο. Ωστόσο, θεωρώ ότι σε τούτη την Επιτροπή μας, που είναι η Επιτροπή Απασχόλησης, δεν είμαστε ΙΜΚΟ, η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μας απασχολεί αλλά μας απασχολεί και η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, η καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ και επομένως ο συνειρμός ο κοινωνικός είναι σημαντικός. Και αυτό το πρόσημο εμείς θέλουμε να γίνει σαφές. Εμείς ως πολιτικοί, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Είμαστε εκλεγμένοι, είμαστε, μας έχουν εκλέξει και αυτή τη δουλειά μας έχουν εκλέξει για να κάνουμε. Και αυτό θέλουμε να δείξουμε στους ε, πολίτες μας. Θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα για μια Ευρώπη κοινωνική. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα στην Ευρώπη. Το πρώτο στοιχείο που αγχώνει τους ε, ε, πολίτες της Ευρώπης είναι η απασχόληση. Και διαρκώς μας ρωτάνε οι πολίτες μας τι κάνει για τη δημιουργία θέσεων, τι κάνει για τις δουλειές μας, για την απασχόληση η Ευρώπη. Και δεν είναι δυνατόν λοιπόν εμείς να κρυφτούμε πίσω από μία ασπίδα, την ασπίδα της ευκολίας και των κοινότοπων λόγων. Πρέπει να πάμε παραπέρα. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Περέρα ίσως σας δυσκολέψουμε λίγο αλλά παρόλα αυτά εμείς θέλουμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Αυτά ήθελα να πω κυρία Πρόεδρε σε όλους, σε εσάς, στους συναδέλφους. Ευχαριστώ φυσικά την Αγνές. Γιατί ξέρετε δεν είναι και τόσο εύκολο να έχουμε μια τόσο αγαστή συνεργασία. Έρχομαστε από δύο διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Θα μπορούσαμε να έχουμε στοιχεία ρήξης. Όχι όμως. Εμείς προτιμήσαμε τη συνένεση, προτιμήσαμε τη συμφωνία και επομένως αυτή η καινούργια φάση που ανοίγεται προβλέπεται λαμπρά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγνιές. Ελίζα Ελίζαμπετ Μοχάν Σαχτιέ. Μεγάλη απόλαυση να σας ακούμε και βεβαίως έχουμε πολλές πολλές ελπίδες. Τούτου λεχθέντος, αρχίζουμε στις 2 με την κυρία Τάισελ, την Επιτροπό και συζήτηση για την κατάσταση στην απασχόληση των νέων. Θα σας ξαναδώ λοιπόν στις 2.